υπάρχουν προβλήματα. Και θα αναφερόμαστε και στη γενική κατάσταση όπως οι συγκεκριμένε υποθέσεις που αναφέρθηκαν στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Για να τελειώσει η συζήτηση να πω πως έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλος της συζήτησης. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη το Αζερμπαϊτζάν η υπόθεση του Ιλγκάρ Μαμάντοφ. Θα δώσω τον λόγο στους συντάκτες για ένα λεπτό η κυρία Γκέγκερ Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Φέτος υποτίθεται πως θα ήταν καλή χρονιά για το Αζερμπαϊτζάν ε, καθώς ε, είχαμε, θα έχουμε και τις εκλογές, αλλά ε, υπάρχει εκφοβισμός της ε, αντιπολίτευσης. Ε. Ο διευθυντής ενός σχολείου του Μπακού και υποψήφιος αντιπολίτευσης, ο κύριος Ιλγκαρ Μαμάντοφ, συνελήφθη. Γεγονό είναι πως το Αζερβαϊτζάν πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις του σύμφωνα με την ΕΣΔΑ. Ειδικά ε, καθώς ε, έρχεται και το 2014 η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, το Αζερβαϊτζάν. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωση του Ιλγκάρ Μαμάντοφ και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων στο Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να εγγυάτε δίκες δίκες για όλους. Σας ευχαριστώ. Χέφνερ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φέτος τον Οκτώβριο ε, έχουν εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν μετά από δεκαετίες διακυβέρνησης της οικογένειας Αλίεφ. Ε, τώρα ο πρόεδρος του κόμματος ε, Δημοκρατική Εναλλακτική Λύση ε, είναι ανθυποψήφιος ε, του κυρίου Αλίεφ. Και μετά από κάποιες διαδηλώσεις στην Ισμαϊλούπολη, μια πόλη πέρα, ε, μετά από τις διαδηλώσεις ε, επισκέφθηκε την πόλη ο κύριος Μαμάντοφ και συνελήφθη για υποκίνηση των διαδηλώσεων στην πόλη στην οποία πήγε μετά από τις διαδηλώσεις. Και αυτή είναι μία μόνο περίπτωση από τις ε, πολλές όπου συναμβάνουν άνθρωποι όχι γιατί έχουν αποδεδειγμένα κάνει κάτι, αλλά γιατί είχαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις από το καθεστώς. Το Αζερβαϊτζάν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς. Αλλά πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως βάση μιας συνεργασίας, βάση μιας συμφωνίας σύνδεσης, πρέπει να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, ελευθερίας των ανθρώπων, αξιοπρέπειας, ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας του συνέρχεστε. Χωρίς σεβασμό για όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία σας ευχαριστώ κύριε Χέφνερ. Για ένα λεπτό κύριε Σχάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Το ίδιο το Αζερβαϊτζάν έχει δεσμευτεί για το σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, του ΟΑΣΕ. Όμως ε, αυτές οι υπογραφές δεν πρέπει να μείνουν μόνο στα έγγραφα. Πρέπει να μεταφραστούν σε πολιτική δράση η καταστολή τη κοινωνία των ΜΜΕ πρέπει να σταματήσει. Ο Έλταρ Μαμάντοφ πρέπει να απελευθερωθεί και να ε, απαλλαχθεί από τις κατηγορίες. Ο εκφοβισμό των δημοσιογράφων, οι πυροβολισμοί κατά δημοσιογράφων, η ε, απαγόρευση ειρηνικών διαδηλώσεων είναι κινήσει. κινήσεις. Ε, καλούμε τον Πρόεδρο Μπαρόσο να θέσει αυτό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανώτατο επίπεδο στις 21 Ιουνίου όταν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αλίεφ. Τα οικονομικά και τα στρατηγικά μα συμφέροντα δεν πρέπει να υπεσκιάζουν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο λαό του Αζερβαϊτζάν κοιτάζει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι είναι μια κοινότητα αξιών και δικαίω. α μην του γυρίσουμε την πλάτη γιατί αξίζουν προστασία των θεμελιωδών του ελευθεριών. Σας ευχαριστούμε κυρία Σάκε. Κάμπνο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι δεν έχω ε, συντάξει το κείμενο. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτό το χαρακτηρισμό από το πίνακα. Για, στο σχέδιο ψηφίσματο θα πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση του Τζερβαϊτζάν να ασχοληθεί με την υπόθεση Μαμάντοφ γρήγορα και με δίκιο τρόπο και θα πρέπει να απελευθερωθεί από τη φυλακή. Ένας υποψήφιος για την Προεδρία δεν θα πρέπει μόνο να μπορεί να θέτει υποψηφιότητα, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξαγάγει και μια προεκλογική εκστρατεία. Στην υπόθεση Μαμάντοφ θα πρέπει να αποφύγουμε αναφορές σε θέματα όπως ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ελεύθερες εκλογές και το γραφείο του ΟΑΣΕ. Έχουμε επιτροπές και αντιπροσωπείες που μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα. Αλλά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται το θέμα αυτό. ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Μπλε κάρτα. Ο κύριος Πόσελτ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν μπορεί να βρεθεί στην δική μας τη θέση. Το 1989 εμείς παλέψαμε για τα δικαιώματα της Πολωνίας και των ε, υπολείπων. Και κάποιοι μας έλεγαν, ε, τώρα μην ασχολείστε, κάντε μυστική διπλωματία. Ευτυχώ δεν το κάναμε, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα. έτσι, Τσάβανο, θέλετε να πείτε κάτι. σε καμία περίπτωση δεν λέω πως δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξεπλάγιν εγώ όταν άκουσα από τον επικεφαλή τη αντιπροσωπείας πως αναβλήθηκαν οι συνομιλίε ε, στον Πακού γιατί κανένας ευρωβουλευτή δεν ήθελε να πάει στον Πακού πλην ενός για να διαπραγματευτεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό αναβλήθηκε το ταξίδι της αντιπροσωπείας. Ένα χρόνο πριν ε, είχαμε ε, συζητήσει, είχαμε επαφές στις Βρυξέλλες. Κανένας ευρωβουλευτής πάλι δεν εμφανίστηκε. Εκεί πέρα πρέπει να συζητάμε τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο για την περίπτωση, με μία μεμονωμένη περίπτωση ενός ανθρώπου. Αυτό είπα εγώ. Σας ευχαριστώ. Κάτι πήγε στραβά εδώ πέρα αγαπητέ συνάδελφε. Ακούγαμε γερμανικά από το αγγλικό κανάλι, πρέπει να το δούμε αυτό. Τον λόγο τώρα τον δίνω στην κυρία Τούρν Χόενστάιν. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, ναι, βεβαίω. Η κυρία Βερζιά, την είχα, είχα διαγράψει ήδη το όνομά σα, ενώ δεν μιλήσατε. Monsieur le Président. Πρόεδρε. Παράξενο που ο κύριος Κανόφ μας λέει ότι δεν είναι συντάκτης του ψηφίσματος και αναγράφεται όμως αυτό στο πίνακα. Τέλος πάντων δεν θα φάω το χρόνο μου με τέτοιες λεπτομέρειες. Πριν από ένα χρόνο εκατοντάδε κατέβηκαν ε, στον δρόμο στον Πακού για να ζητήσουν δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Ε, ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, σχήμα καταστολής. Ε, όλοι οι αντιρρησίε, όλοι οι διαδηλωτέ πετάχτηκαν μέσα στη φυλακή, εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του τύπου που του εκπροσώπησαν Επίση υφίστα την ίδια καταστολή αυταρχικός ε, πρόεδρος ε, Αλίεφ ε, δεν σταματάει εδώ και χρόνια να προβαίνει σε αυτές τις πολιτικές κρατήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από δύο μήνες οι αρχές του Αζερβαϊτζάν χρησιμοποίησαν σφαίρες με καουτσού και δακρυγόνα, ακριβώς αυτά που καταγγέλουμε σε άλλες χώρες. Από το 89 και μετά αυτά συμβαίνουν. έχουμε από το 99 μια εταιρική σχέση σχέση. Ανήκει στην ανατολική εταιρική σχέση του Αζερβαϊτζάν και ε, διαπραγματευόμαστε τώρα μία ε, συμφωνία σύνδεση. Εσεί διαπραγματεύεστε, για να είμαι ακριβή. Ε, τι μαθήματα μπορούμε να λύσουμε από την παρελθούσα εμπειρία, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε κατά το ελάχιστο να επικρατήσει ένα κράτο δίκαιο, τι απαιτούμε από αυτού. Α μάθουμε από το παρελθόν επιτέλου. Τέτοιε διαπραγματεύσει για συμφωνία σύνδεση υπήρξαν και με την Τινησία του Μπέναλη. Ε, και δεν έχουν πλέον κανένα νόημα αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ε, κύριε Λεβαντόσκι, δώστε μας μια απάντηση. Σας παρακαλούμε πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούνοντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την σύλληψη κάποιων ε, πολιτικών αντιπάλων που θα μπορούσαν ε, να, γίνουν ε, πρόεδροι έτσι κάποια στιγμή. Είναι σκανδαλώδες. Ειδικά σε χώρες οι οποίες θέλουν να αποδείξουν πως έχουν δημοκρατικά θεσμικά όργανα. και θα αναλάβουν μάλιστα και την Προεδρία την εναλλασσόμενη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε πως υπάρχει και η συμφωνία σύνδεσης ε, και μέσα σε όλα αυτά μπαίνει η αντιπολίτευση στη φυλακή. Κοιτάξτε, σε όλες τις ε, συζητήσεις και σε όλα τα θέματα που είχαμε ε, κάποιες σκληρότερες απόψεις. Είχαμε και πιο σκληρές φωνές για την περίπτωση Μαμάντοφ. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε και τώρα. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητές ονόματος των ομάδων. Η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταδικάζω τη σύλληψη του Ιλγκα Μαμάντοφ στις 4 Φεβρουαρίου που έγινε μετά από ειρηνικές διαδηλώσεις δεν δόθηκαν λόγοι για τη σύλληψη και τη φυλάκισή του. Ψευδείς κατηγορίες απαγγέλθησαν κατά του Ίγκαρ Μαμάλντοφ. Κατηγορείται για κάποιο είδους βίαιη δράση. Οι διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικές. Και οποιοδήποτε λαός θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κρίνει την κυβέρνησή του. Το άκρο νάτων της ηρωνίας είναι ότι ο Έλγκαρ Μαμάντοφ δεν ήταν καν παρόν στις διαδηλώσεις. Παραμένει γεγονός Ο Ίγκα Μαμάντοφ λοιπόν έχει φυλακιστεί και έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του. Είδαμε παρόμοια πράγματα να συμβαίνουν στην Τουρκία και στη Ρωσία. Θα πρέπει να πολεμήσουμε για τη δημοκρατία, να πολεμάμε καθημερινά. Ευχαριστώ κυρία Μάκοβαϊ. Για ένα λεπτό η κυρία Σενίσιν. Με μικρόφωνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Αζερβαϊτζάν έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να ασχολείται όμως, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα των πολιτικών κρατουμένων. Δεν, έχει ελευθερο, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία. Το διαδίκτυο είναι περιορισμένο και τίθενται περιορισμοί στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και δεν υπάρχει ελευθερία στον αφορά δηλώσει. Καλούμε τις αρχές της χώρας να αφήσουν τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ να λειτουργήσουν με ασφάλεια και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ζωτική σημασία για την ε, δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Είναι κρίσιμο θέμα για την συμφωνία σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της συνελεύσεως και όλα αυτά τα θέματα. Ο πρόεδρος Μπαρόσο πρέπει να τα θέσει τα ζητήματα όταν ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν επισκεφτεί τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πω ότι έκανα κάποιες, κάποιους υπολογισμούς. 32 από εμά βρισκόμαστε στην αίθουσα της Ολομελίας. Και θα ζητούσα την κυρία Τούν Φον να μην ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τις απόψεις εκείνων που δεν είναι στην αίθουσα της Ολομέλειας. Δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει. Και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους απουσιάζουν μέλη του Κοινοβουλίου από την Ολομέλεια. Οι παρόντες δεν πρέπει να διατηνόμεθα έναντι των φορολογουμένων ότι ε, είναι 750 από εμά παρόντες στην αίθουσα. Είμαστε μόνο 32 στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Η κυρία Βερζιά από την ε, αριστερά δεν θα πρέπει να επικρίνει την ομάδα τη δική μου και τον κύριο Τζάμπερνοχ. Η ομάδα της κυρίας Βερζιά έχει μιλήσει με πολλές γλώσσες και με πολλές προσεγγίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιες από τις χώρες μας κατά το παρελθόν. Έχουμε μπλε κάρτα από τον κύριο Χέφνερ. Κύριε Τσαρνέτσκι, Θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Χέφνερ. Κύριε Χέφνερ. Κύριε Τσαρνέσκη, αντιλαμβάνομαι πως ε, θέλετε να φύγετε αμέσως μετά από αυτά τα οποία είπατε. Αλλά πριν πάτε για άλλες δουλειέ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το οποίο είπατε. Ε, δεν ξέρω. Δεν έχετε καταλάβει τους κανόνες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εδώ πέρα βρίσκονται βουλευτές Και εδώ πέρα είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων. Και σας παρακαλώ να μην επιτίθεστε στους ανθρώπους που κάνουν εδώ πέρα αυτή τη δύσκολη δουλειά. Αντί να ασχολούνται με τις υποθέσεις άλλων χωρών. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαρνίσκη και η κυρία Βεζιά θα ήθελα να σας κάνει μια ερώτηση. Μπορείτε να ακούσετε και αυτή την ερώτηση και να δώσετε μια απάντηση. Κύριε Βεζιά. Δεν ξέρω αν είναι μπλε κάρτα ή κάτι προσωπικό μου. Απλώς εγώ θέλω να αντιδράσω σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, που ε, ξεπλάγει γιατί αναγράφεται ο συντάκτης. Να τα βάλει με τους συναδέλφους, το έχει με το κοινοβούλιο. Για την πολιτική το ομάδα δεν είπα τίποτα άλλο. Σε σχέση με τις διαφορές ανάμεσα πολιτικές ομάδες, ε, για τακτοποιήστε τα ενίκο πρωτού αρχίζετε να επιτίθεστε σε άλλους. Ευχαριστούμε. Στανέσκι. Ευχαριστώ. Μου φαίνεται ότι ο κύριος ε, Χέφνερ ε, ηθελημένα ε, δεν αντελήφθη το τι είπα νωρίτερα. Εγώ είπα ότι οφείλουμε σεβασμό προς τους 32 παρόντες ε, βουλευτές και ότι δεν ενδείκνυται να αναφερόμαστε σε βουλευτές που για οποιοδήποτε λόγο αποσιάζουν. Κυρία Βεργιά, δεν αναφερόμουν στο ψήφισμα εγώ αναφερόμαι στι απόψεις της δικής σας πολιτικής ομάδας στα πλαίσια άλλων συζητήσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσαρνέτσκι. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Τσιόμπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το Αζερμπαϊτζάν είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Ο αγωγός Ναμπούκο και το πρόγραμμα Ναμπούκο, εάν τελικά υλοποιηθεί, θα κάνει πολλά για, την, για τον ασφαλή εφοδιασμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ενέργεια. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με την εν λόγω χώρα και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Και αυτό είναι το βασικό θέμα. Παρά κάποιες αναλαμπές ελπίδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν, το πρόγραμμα των εκλογών έχει δείξει ότι ίσως απογοητευτεί ο υπόλοιπος κόσμος εάν θεωρούσε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήταν ένα, μια μονάδα μέτρηση για τη σχέση μεταξύ χωρών. Οι προεδρικές ε, εκλογές του Οκτωβρίου ε, θα καταφτάσουν και είναι φυλακισμένος ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Αυτό δείχνει ότι ο πρόεδρος Αλίεφ δεν είναι και ο μεγαλύτερος δημοκράτης στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί. Νομίζω ότι αυτές οι απόψεις θα πρέπει να ακουστούν και νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι λόγοι αυτοί προς σωστή κατεύθυνση. Είναι πράγματα που θα πρέπει να λέμε δυνατά και καθαρά. Θα πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θέλουμε το Τζερμπαϊτζάν να πέσει στα χέρια στην αγκαλιά της Ρωσίας που περιμένει. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Ξεκινάει ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, η Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν έχουν πολλά κοινά, ειδικά όσον αφορά την περιφρόνηση για την ελευθερία του τύπου, την ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε και την δυσανεξία στην αντιπολίτευση. Και αναμέναν πάρα πολλά από τις εκλογές στο Αζερβαϊτζάν ε, τον Οκτώβριο. Ε, τελικά τα πράγματα ε, εξελίσσονται απογοητευτικά. Και η περίπτωση Μαμάντοφ είναι χαρακτηριστική. Υποψήφιος πρόεδρος φυλακίζεται με ψευδείς κατηγορίες της υποκίνησης ταραχών. Ε, αναβάλλεται δύο φορές η δίκη και κρατήτε Και θα τον δικάσουν ή απελευθερώσουν μετά τις εκλογές από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να απελευθερωθεί το στομότερο δυνατόν, για να είναι δίκαιες οι εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον βασικό. Σας ευχαριστώ. Κρετού για ένα λεπτό. Συμφωνώ με όσους διαφωνούν με τη μεταχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς των αρχών του Αζερβαϊτζάν. Είναι όντως απογοητευτικά τα όσα συνέβησαν, κυρίως επειδή θα έχει αναλάβει την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Αζερβαϊτζάν το 2014. Ο Ήλγαρ Μαμάντοφ, ο προεδρικός ανθυποψήφιος, ε, δίωκεται. Αυτό δείχνει επιδείνωση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Θα έπρεπε η χώρα αυτή να οργανώσει δημοκρατική εκλογική αναμέτρηση, να σέβεται την αντιπολίτευση και να μην ποινικοποιεί δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Καλό τον πρόεδρο Μπαρόσο να μεριμνήσει ώστε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα από άλλες χώρες. Θα πρέπει ε, να θέσετε αυτό το ζήτημα με τις αρχές του ε, Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικός περιφερειακός φορέας είναι βασικός εμπορικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ενώσεω και ας ελπίσουμε ότι η σημασία της χώρας θα αυξηθεί, κυρίως όσον αφορά τον εφοδιασμό τον ενεργειακό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τα κάνουμε τα πράγματα εύκολα για το Ετζερμπαϊτζάν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητούμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έναν άλλον εταίρο και πρέπει να ζητήσουμε και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από ένα πραγματικό εταίρο, το Τζερμπαϊτζάν Θα ήταν κακό να παρεξηγηθεί ο κ. Τσάμπαρνοχ. Ο κ. Τζάμπαρνοχ ηγείται τη αντιπροσωπεία που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και αν επέκρινε οποιονδήποτε, επέκρινε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας που δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της διότι οι ευρωβουλευτές δεν εμφανίζονται στις συνεδριάσεις. Το ECR είναι σαφές από αυτού του θέματος και έχουμε υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία και Να σας παρακαλέσω όλους. Ε, έχουμε τέσσερις που έχουν ζητήσει το λόγο, πέντε και δύο λεπτά μόνο. Πρέπει να μείνετε στο ένα λεπτό ο καθένας. Ε, κυρία Σαγιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μαμάντοφ είναι πολιτικός αντιπολίτευσης, ο οποίος ε, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ε, για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και πολύ καιρό. Το Φεβρουάριο συνελήφθη σε μια ειρηνική διαδήλωση και τώρα αντιμετωπίζει πλαστές ε, κατηγορίες η Human Rights Watch ε, ζήτησε από το Αζερβαϊτζάν, την κυβέρνηση δηλαδή, ε, να απαγγείλει ε, κατηγορίες στον κύριο Μαμάντοφ γιατί θα γίνει και θα αναλάβει και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης το Αζερβαϊτζάν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Όγιλοντ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σαν στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Αζερβαϊτζάν γνωρίζει και ακολουθεί θρησκευτική ανοχή και κοσμικό κράτο είναι και σέβεται και κάποιου κανόνες οικονομικούς και οι εταίροι μα στο Αζερβαϊτζάν περιμένουν πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ψήφισμα υποστηρίζει τι συνεχιζόμενε διαπραγματεύσει για την Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν. Ταυτόχρονα αυτό το ψήφισμα μα υπενθυμίζει και υπενθυμίζει στου φίλου του Αζερβαϊτζάν ότι είναι μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη με όλε τι υποχρεώσει περί δημοκρατία, κράτου δικαίου και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και καλό τον να συνεχιστεί ο ανοιχτό και καλό διάλογο που λαμβάνει η χώρα με τη δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν για να συμβάλλουμε στην προσέγγιση των δύο λαών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Αζερμπαϊτζάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το, τη συζήτηση, θα έλεγα ότι είναι δυσανάλογη επιτιθέμεθα κατά του Αζερβαϊτζάν αλλά η συζήτηση για τη Ρωσία ήταν υπιότερη. Ε, Ήμασταν πολύ ήπιοι εναντί της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Στη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρουμε την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης. Η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, παραβιάζει την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης. κατασκεύασαν αγωγό αερίου που, κάτω από τη Βαλτική που συνδέεται με τη Ρωσία. Και πληρώνουν τεράστια ποσά στους Ρώσους. Μεγάλες συμφωνίες επιχειρηματικές έκανε η Γερμανία με τη Ρωσία πίσω από την πλάτη της Πολωνίας. Πρέπει να μιλήσουμε για τους Μαγνέσκι και Κοντακόφσκι. Αλλά και πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί και για τα άλλα θέματα γενικά. Ευχαριστώ κύριε Κόσκι. Η κυρία Κορχόλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχει αναλάβει δέσμευση το Αζερβαϊτζάν ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέραν αυτού, αναμένεται να αναλάβει το 2014 την ε, Προεδρία Εκπεριτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όμως, μετά τη σύλληψη του Ιλντερ Μαμάντοφ, που ηγήθηκε της αντιπολίτευσης ε, στην εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε την αποφυλάκησή του ε, και την δίκαιη δίκη που αξίζει. Όπως και σε προηγούμενα ψηφίσματα για το Αζερβαϊτζάν, ε, όντως πρέπει να αναφερθούμε στην ελευθερία για τα ΜΜΕ, είναι κατακριτέα η παρενόχληση δημοσιογράφων, υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να κάνει τα δέοντα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστούμε κυρία Κόρχολα Χίπνορ για να κλείσει η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λαμβάνω το λόγο για το Αζερβαϊτζάν, άλλη μια χώρα που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διώκει ανθρώπους που έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Αυτή τη φορά μιλάμε για τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ, υποψήφιο για πρόεδρο, υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Τον φυλακίζουν σαν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να ήταν δολοφόνος. Πρόκειται όμως για πολιτικό της αντιπολίτευσης. Η σύλληψη Μαμάντοφ ε, που ήταν πίσω από πολλές δημοκρατικές πρωτοβουλίες οδήγησε σε ανησυχία στο Αζερβαϊτζάν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Αρχές Μαΐου ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης από τις ζερικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς ε, κρατούμενους, αλλά εις ότα μία κόντων έπεσε η έκκληση ε, κάτι πραγματικά αποκοστικό, ειδικά σκεφτόμουν του έξι μήνε, αναλαμβάνει το Αζερβαϊτζάν την Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ πέρα η διαδικασία και τώρα θα ακούσουμε από την Κομισιόν τον κύριο Λεβαντόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, και πάλι θα μιλήσω εκπροσωπώντας την ε, Βαρόνια Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Σημεία τα όσα είπατε. Η περίπτωση Μαμάντοφ είναι σοβαρή, αξίζει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρώτον λόγω του τρόπου χειρισμού και δεύτερον λόγω της σημασίας που έχει βεβαίως η δυνατότητα η αντιπολίτευση να κινείται ελεύθερα. Ε, ε, σε μια προεκλογική περίοδο. Και ανησυχούμε για την κράτηση του κυρίου Μαμάντοφ στην απομόνωση, όπου δεν μπορεί να τον επισκεφτεί ούτε η οικογένειά του, ούτε φαΐ δεν μπορεί να λάβει εκτός φυλακής. Και, γενικότερα, ε, και προφανές η κράτησή του βεβαίως δεν του επιτρέπει να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως και η υπατή εκπρόσωπος ε, και ο επίτροπος ο κύριος Φίλε παρακολουθούν στενά τις ε, πολιτικές εξελίξεις και στις ε, συναντήσεις τους με την ηγεσία του Αζερβαϊτζάν και σε δύο πολύ έντονες δημόσιες δηλώσεις ζήτησαν ανεξάρτητη και διάφνη έρευνα και πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν σιωπούν. Ναι, ναι και αυτό βεβαίως ε, είναι σύμφωνο με τις αρχές ε, της δημοκρατίας ε, στον ευρωπαϊκό χώρο. Κάτι το οποίο δεν λαμβάνει μόνο τις τυπικές προϋποθέσεις των εκλογών αλλά και τις ελευθερίες των πολιτών να μπορούν να συνέρχονται, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδικτύο. Οπότε συζητήθηκε και το ζήτημα της δικαιοσύνης και του πώς λειτουργεί και όχι μόνο η περίπτωση Μαμάντοφ και βεβαίως αυτό επίσης είναι μέρος του διαλόγου με το Αζερβαϊτζάν όπως επίσης αναφέρθηκε πρόκειται για έναν εταίρο πολύ σημαντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η σχέση μας νομίζω θα πρέπει να μας επιτρέπει να μιλάμε ε, ειλικρινά όταν αυτό χρειάζεται. Και νομίζω είμαστε σε αυτή την εποχή και σε αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ληφθεί υπόψη και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα όπως το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, η νομοθεσία περί δυσφήμισης και η εκλογική νομοθεσία, αλλά σας διαβεβαιώ πως αυτό τα οποία συμβαίνουν στο Αζερβαϊτζάν τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και έχει κινητοποιηθεί η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας συναντήθηκε με τον κύριο Μαμάντοφ στις 4 Απριλίου. Είναι σε στενή επαφή με την οικογένεια και τους δικηγόρους του κυρίου Μαμάντοφ και αυτό αφορά όχι μόνο τον κύριο Μαμάντοφ αλλά και τους άλλους κρατούμενους, ο κύριος Τόφικ Γιακούμπλου, ο οποίος επίσης ε, είναι προφυλακισμένος και μπορώ να σας πω πως η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκε τον κύριο Γιακούμπλου στην φυλακή και όπως και στην περίπτωση Μαμάντοφ συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε ε, σε όλες τις ε, σχετικές ε, περιπτώσεις και παρακολουθούμε όπως είπα αυτές τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Έχουν κατατεθεί έξι ε, προτάσεις ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη το θέμα για την